Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε καθυστερήσει. Ε, να περιμένουμε όλους να εγκατασταθούν. Παρακαλώ καθίστε. Δύο είναι τα σημεία στην ημερήσια διάταξη μέχρι και τις 4.30 και διότι τότε θα ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Λοιπόν, καταρχάς, θα εξετάσουμε μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για το κοινό σύστημα φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ο κύριος Ίγκλη είναι ο εισηγητής και ο Όδης είναι ο κύριος Κοριαρίντε Κάμπος, Μάντος. Κάμφε, κύριε Κάμφερ, μιλάτε εξ ονόματος των Πρασίνων ή όχι. Ή, ενδεχομένως, ναι. Και ο κύριος Ντε βεβαίως. Ε, εκ μέρου της ομάδας μου δεν ξέρω ποιο θα τοποθετηθεί, ίσω εγώ. Λοιπόν, ας ε, ξεκινήσουμε λοιπόν. Υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Ναι, εσείς, κύριε Ντίμερ. Καλώς. Κύριε Άγγλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων σήμερα για το θέμα. κατ' θα μιλήσω αγγλικά γιατί τα έγγραφα που μου δόθηκαν ήταν στα αγγλικά οπότε ε, θα μιλήσω και αγγλικά να τονίσω μερικά βασικά θέματα για τη συζήτηση τα οποία νομίζω ότι έχουν σημασία πρώτα πρώτα θα μιλήσω για το FTT είναι ο φόρος αυτός Financial Transaction Tax ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε πού επιβάλλεται ο φόρος αυτός στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές αυτές καθεαυτές. Δηλαδή τις συναλλαγές που κάνουμε όλοι στην ιδιωτική μας τη ζωή αλλά και καταναλωτική πίστη και τα και τα λοιπά. Γιατί φτιάχνουμε τη γνωμοδότηση, γιατί θεωρούμε ότι το ζήτημα αυτό σχετίζεται με τη λειτουργία της ε, εσωτερικής, ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Um, Η Κομισιόν επισύναψε στην πρότασή της και μία μελέτη αντικτύπου που λέει ότι, ότι το προϊόν αν θέλετε της πρώτες αυτής δηλαδή το έσοδο θα είναι 57 δις ευρώ περίπου θα επηρεαστεί θετικά και η ανάπτυξη κατά το ίδιο ποσό περίπου δηλαδή από τη μια θα χάσουμε, θα περάσει αρνητικά με συγχωρείτε την ανάπτυξη. Απ' τη μια λοιπόν θα χάσουμε ένα ποσό, αλλά θα, απ' την άλλη μεριά θα πάρουμε περίπου το ίδιο ποσό. Βεβαίως θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω το κατά πόσο θα ήταν λογικό να υπολογιστεί και τι θα γινόταν αν οι συντελεστές ήταν τελείως διαφορετικοί. Δηλαδή, ίσως θα χάναμε περισσότερα από την ανάπτυξη, από τα έσοδα που θα κάναμε. Τέλος πάντων, 0,1% είναι ο συντελεστής ε, που προτείνει η Κομισιόν για τις συναλλαγές. Γενικά 0,01% για τα παράγωγα. Υπολογίζεται ότι οι εμπορικές συναλλαγές, μπορεί να, οι μπορούν να πέσουν 70% μετά την επιβολή του φόρου αλλά και για ιδιαίτερα μεγάλες συναλλαγές ενδεχομένως να πέσουν αυτές κατά 90%. Άρα, κατά τη δική μου την άποψη, θα έπρεπε να πούμε ότι θα χαθούν συναλλαγές κατά 90% τουλάχιστον για τα παράγωγα και άλλες μεγάλες συναλλαγές αυτό έχει μεγάλη πολιτική σημασία και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οπότε ενδεχομένως θα πρέπει να αλλάξουμε τους συντελεστές. Θα πρέπει να υπολογίσουμε ποιο, τι επίπεδο συναλλαγών, όγκο συναλλαγών θέλουμε να έχουμε στην εσωτερική αγορά για να δούμε πώς μας βολεύει να κινηθούμε. Από εκεί και πέρα, η ΔΕΒΕ και η Επιτροπή Ανάπτυξη και η Επιτροπή Προπολογισμών θα κάνουν τις δικές τους γνωμοδοτήσεις. Βεβαίως, κατά πάσα πιθανότητα, η Επιτροπή Ανάπτυξης θα πρέπει, μάλλον θα πει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί θέλουμε να υπάρχουν κονδύλια για να μπορούν να, διατη, να διατεθούν για αναπτυξιακούς σκοπούς ε, Υποθέτω βέβαια ότι θα το πει αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα για την Επιτροπή Προπολογισμού δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει ο φόρος αυτός τον προϋπολογισμό. Ίσως η Επιτροπή Προϋπολογισμού θα πει ότι είναι μη πόρος αυτός, non-resource, για να μην επηρεάσει το προϋπολογισμό. και θα, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να παραμείνει μη πόρος αυτός ο φόρος, τα έσοδα από το φόρο αυτό. Τώρα, βεβαίως η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων έχει ασχοληθεί με το θέμα και βάσει της δουλειάς που έγινε νομίζω ότι τελικά θα αποφασιστεί ότι ο φόρος αυτός δεν θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά μόνο στην Ευρωζώνη. Δεν το έβγαλε από το κεφάλι της βέβαια η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Αυτό παίζει εκεί ρόλο η Γαλλία και η Γερμανία. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει εσωτερική αγορά της Ευρωζώνης. Μόνο εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι το πιο σημαντικό πρέπει να προσέξουμε εδώ είναι ότι θα πρέπει ο φόρος να επιβληθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι σε ένα χώρο μικρό, σε ένα χώρο μικρότερο του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή στην Ευρωζώνη θα πρέπει να προσέξουμε να μην ε, επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της ιστορικής αγοράς ο φόρος αυτός δηλαδή τελικά θα έλεγα ότι δυο πράγματα είναι σημαντικά πρώτον πού θα επιβληθεί ο φόρος αυτός Δεύτερον, ποιος θα είναι ο δίκτυπος της φορολογίας αυτής σε κάποιες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και εμπορικών συναλλαγών, μήπως θα πρέπει να υπάρξουν εδώ και άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις για να μην ε, ξεφύγει τον πλήρη έλεγχο η κατάσταση αυτή. Αυτά λοιπόν σαν πρώτες σκέψεις από πλευράς μου και περιμένω τώρα να ακούσω τις δικές σας απόψεις. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Σαφέστατη η παρέμβασή σας δημιουργεί ένα πλαίσιο με το οποίο θα συζητήσουμε. Ο καθηγητής Κορίρα Κάμπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πρώτα πρώτα τον εισηγητή για την ε, πολύ καλή και ευαίσθητη θα έλεγα εισαγωγή την οποία μας έκανε. Παρουσιάζει τα πράγματα απλά. Τα παρουσιάζει απλά, αλλά τα πράγματα είναι περίπλοκα. Η χρηματοπιστωτική κρίση, μάλλον η κρίση, η οικονομική κρίση στην Ευρώπη οφείλεται εμπολίσει το χρηματοπιστωτικό τομέα και η πρόταση αυτή προσπαθεί να ξεκινήσει μία η κίνηση εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα επηρεάσει όλο τον κόσμο. Τα πράγματα όμως είναι περίπλοκα και βλέπουμε ότι όλοι δεν συμφωνούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αντιρρήσεις. Γι' αυτό λένε κάποιοι θα πρέπει να εφαρμοστεί ο φόρος αυτός μόνο στην Ευρωζώνη. Αλλά επειδή μιλάμε ουσιαστικά εδώ για παγκόσμια συνεργασία, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν θα έπρεπε να γίνει. Το γιατί πρέπει να επιβληθεί ο φόρος αυτός και με τους συντελεστές που προτείνονται. Εξηγείται στην πρόταση. Αλλά ε, ο, το χρηματοπιστωτικός τομέας είναι μάλλον ρευστός αν θέλετε. Μάλλον ένας τομέας με ιδιαίτερα ψηλή κινητικότητα και η εφαρμογή σε ένα μέρος του κόσμου ενδεχομένως να οδηγήσει κάποιους οργανισμούς ε, χρηματοπιστωτικούς να μετακινηθούν. αυτά είναι γνωστά και ε, ε, υπάρχουν άποψη, υπάρχουν πολλοί που είναι αντίθετοι προς την πρόταση που την, ε, το υποστηρίζουν, ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Από την άλλη μεριά υπάρχουν τα επιχειρήματα αυτών, των, που υποστηρίζουν την πρόταση ζητούνται από κάποιους εξαιρέσεις εξαίρεση λόγω χάνει των κεντρικών τραπεζών αλλά εξαιρέσεις είναι επικίνδυνες και μπορεί τελικά να οδηγήσουν και σε μια ανεξέλεκτη κατάσταση και ε, απώλεια ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ή όσον αφορά τώρα την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας μέσω τέτοιου είδους μέτρων δεν ε, είμαστε και 100% σίγουροι ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Πιστεύουμε ότι ο αντίκτυπος του φόρου αυτού θα επηρεάσει όλους τους τομείς της οικονομίας και βεβαίως το εργαλείο αυτό θα εφαρμοστεί μόνο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε πώς θα επηρεαστούν και οι εταιρείε και τα νοικοκυριά από το φόρο αυτό. Από εκεί και πέρα Πώς, τι θα κάνουν οι εταιρείε, θα μπορέσουν να μετακυλήσουν το επιπλέον αυτό κόστος του φόρου. Αυτό θα ήταν αντίθετο με το σκοπό που ε, επιδιώκουμε εδώ, που ζητούμε δηλαδή από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τις τράπεζες να συμμετάσχουν στην αντιμετώπιση της κρίσης, να συμβάλλουν και αυτές. Ε, αν, αυξήσουν, αν η αύξηση του κόστου των τραπεζών ε, επηρεάσει όλη την οικονομία, εταιρείε και νοικοκυριά, αυτό θα είναι γενικώ αρνητικό. Αν όμω δεν μπορέσει να μετακυλιστεί το κόστο, τότε ενδεχομένως να επηρεαστούν μόνο οι ισολογισμοί των εταιριών και θα πρέπει να το προσέξουμε και αυτό. Τώρα, το τα έσοδα εδώ που υπολογίζονται όπως ακούσαμε ως έσοδα από το φόρο αυτό θα πρέπει να τα δούμε με κάποιο σκεπτικισμό δίνεται μια μεγάλη γκάμα βέβαια για το, τα έσοδα που σημαίνει ότι κανείς δεν είναι σίγουρος για το τι θα γίνει και βεβαίως λέγεται ότι να τα έσοδα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να μην επιβαρύνουν ιδιαίτερα να χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν ε, συνεισφορές, εισφορές των κρατών μελών που θα έπρεπε να αυξηθούν αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο άρα το όλο, το, η όλη υπόθεση είναι αρκετά ασαφής κατά την άποψή μου Μάντερς Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. άκουσα την αγγλοσαξονική προσέγγιση του εισηγητή. Μ' άρεσε. Και συμφωνώ πολύ με αυτά που είπε. Γιατί λέω γιατί να επιβάλλουμε έναν επιπλέον φόρο τη σήμερα ημέρα. Τι είναι, είναι η επιπλέον ίδιο σπόρος επειδή είμαστε 27. Από την άλλη μεριά Μήπως το κάνουμε για να αποφευχθούν ε, ε, έξτρα χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που δεν χρειάζονται να γίνουν. Ναι, ωραία. Αλλά τότε κάποιες συναλλαγές θα τις φορολογούμε, κάποιες όχι. Αν κάνουμε κάτι τέτοιο, ίσως θα καταστούν διαφανέστερες οι συναλλαγές, οι χρηματοπιστωτικές που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη. Αυτά είναι σοβαρά ερωτηματικά που πρέπει να απαντηθούν. Χτες ο Επιτρόπος ανακοίνωσε μια νέα μελέτη αντικτύπου για το θέμα τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε και άλλες αναβολές γιατί περιμένουμε μπας, μήπως γίνει και άλλη μελέτη αντικτύπου ή να γνωρίσουμε τι λέγεται στην καινούργια μελέτη είναι σίγουρα τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Εγώ πάντως αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να υποστηρίξω την ιδέα. Έχω και εγώ τις αμφιβολίες μου, σαν και αυτές που ακούσατε από τους προηγούμενους ομιλητές. Καλό θα ήταν να ξέρουμε τι θα κοστίσει αυτή η υπόθεση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και να ξέρουμε και πόσες συναλλαγές θα βγουν και θα λαμβάνουν χώρα εκτός Ευρώπης και πόσα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα καταλήψουν την Ευρώπη. Θα πρότεινα λοιπόν να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μετά την μελέτη αντικτύπου, την καινούρια που θα φτιάξει η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εμίλη, θέλεις να πάρεις το λόγο? Παρακαλώ. Ναι. Δεν είμαι σκιώδης εισηγήτρια. Ο Πασκάλ Καμφά είναι ο σκιώδης εισηγητής. Και θα τον δείτε βέβαια κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μπορώ όμως να τοποθετηθώ εκ μέρους της ομάδας μου αρκετά καλά πιστεύω. Να πω ότι σε γενικές γραμμές διακύμεθα πολύ ευμενώς σε έναν ευρωπαϊκό ε, φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή χρηματιστηριακών συναλλαγών. Για λόγους δικαιοσύνης καταρχάς είναι ο πιο βασικός λόγος. Θα πρέπει ο κλάδος αυτός να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση των ευρωπαϊκών οικονομιών. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο έχει ένα θετικό κανονιστικό αποτέλεσμα, ρυθμιστικό αποτέλεσμα. Πρέπει να δούμε ποιος θα το πληρώνει. Θα το πληρώνει ο, όποιος κάνει ε, trading, ε, χρηματιστηριακές συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρηματιστηριακές συναλλαγές υψηλής συχνότητας μέσω υπολογιστών ε, πάρα πολλές αναδευτερόλεπτο αγοραπολισίες, αναδευτερόλεπτο και εν μέρη ευθύνονται και για την πρόκληση της κρίσης. Νομίζω λοιπόν ότι ρυθμίζεται αυτό το κομμάτι του χρηματοπιστωτικού τομέα, ο, χρηματο, ο χρηματιστηριακός δηλαδή ε, ε, υποκλάδος και βεβαίως κατά τρίτο λόγο μπορεί να μας αποφέρει και έσοδα. Εξαρτάται πώς θα σχεδιαστεί και τι έσοδα θα αποφέρει και πώς, πόσο τα έσοδα αυτά θα είναι υψηλότερα από τις απώλειες σε επίπεδο εθνικού ΑΕΠΕ λόγω της θέσπισης αυτής της φορολόγησης και κατά τέταρτο λόγο θα ενισχύσει την ανάπτυξη και τις, τις θέσεις απασχόλησης. Λέγεται ότι θα επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης, αλλά να αναλογιστούμε τι είδους θέσεις απασχόλησης θέλουμε και τι είδους ανάπτυξη θέλουμε. Λόγω της κρίσης έχουν χαθεί 9 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι θέσεις απασχόλησης βεβαίως με νοιάζουν, αλλά χρειαζόμαστε αηφορία στον, ε, στην οικονομία μας. Και αν πρέπει να συρρυκνηθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας στο μέλλον για να παραμείνει αηφόρος, ε, τότε αυτό δεν θα με πειράζει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή ήδη οι πόροι, τα έσοδα αυτά ή να επιστραφούν ε, στις εθνικές κυβερνήσεις. Φανταζόμαστε όλοι ποια θα είναι η τοποθέτηση η δική μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βεβαίως, αλλά και από την άλλη πλευρά των κρατών. Βεβαίως ως πράσινοι εμείς είμαστε υπέρ των ε, ευρωπαϊκών ίδιων πόρων. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Νομίζω ότι όλοι οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αυτή τη στιγμή ε, επιδιώκουν την ε, συλλογή των φόρων και από τη στιγμή που θα υπάρξει νέος φόρος θα θελήσουν πάρα πολύ να τον καρποθούν. Δηλαδή αν θέλετε να, έχουν, ε, να υπάρχει εθνική αρμοδιότητα για το θέμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρουσίασε μια σαφή πρόταση. Ε, είναι κάπως ελληματική, έχει κάποια μειονεκτήματα θα πρέπει να συζητήσουμε το σχεδιασμό αυτής της πρότασης, όχι τόσο το υπέρ ή κατά, ναι ή όχι σε ένα τέτοιο είδους φόρο, αλλά να διασφαλίσουμε ότι θα είναι ένα μοντέλο εμπνευσμένο από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα ισχύει συνολικά για όλες τις εταιρείες τις ε, ε, εισηγμένες. Αυτό θα σημαίνει ότι και οι ξένες εταιρείες θα ε, συνεισφέρουν φορολογικά πολλές άλλωστε από τις ε, εταιρείες που φορολογούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο βλέπουν ουσιαστικά τους φόρους τους να πληρώνονται από άλλες εταιρείες που δεν ανήκουν στο City του Λονδίνου. Ε, παρόλα αυτά το City του Λονδίνου δεν έχει καθόλου συρρυκνωθεί. Το λέω αυτό για να πω ότι εάν σχεδιάσουμε το σύστημα σωστά ε, δεν θα υπάρχει ε, πρόβλημα. Ε, το σουηδικό μοντέλο έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι λειτουργικό. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πολύ το σχεδιασμό. Επιπροσθέτως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την άποψη των ε, καταναλωτών. Κάποιοι πιστεύουν ότι αν υπάρχουν επιπρόσθετοι φόροι, τότε τελικά θα μετακυλιστούν στον καταναλωτή, ο οποίος και θα τους αναλάβει στη τελική. Ε, απαντούμε σε αυτό λέγοντας ότι ναι, ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος, αλλά οφείλουμε να αυξήσουμε τη διαφάνεια στο τραπεζικό κλάδο και να γνωρίζουν περισσότερο οι καταναλωτές τι ακριβώς γίνεται. Άλλωστε, αν ε, υπάρχει, αν θέλετε, μια συστημική τάση μετακύλησης του βάρους προς τον καταναλωτή, ενδεχομένως μπορούμε να αναλάβουμε δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ξέρω τι ε, μπορεί να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί είναι ελεύθερη αγορά και ελεύθερη ο καθορισμός των τιμών. Αν όμως συστηματικά πλήττεται το καταναλωτής και καλείται να φέρει ο ίδιος το βάρος αυτό, ίσως ενδεχομένως να έχουμε περιθώρια δράσης. Και ως προς το χρονοδιάγραμμα η λέξη είναι τώρα, για να εμπνεύσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει καλύτερη δουλειά. Είναι ε, η κατάλληλη χρονική στιγμή να παρέμβουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ο Ντένις Τεγιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω τα εξής που ε, μου ήρθαν έτσι αυθόρμητα στο μυαλό. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερω η τεχνική στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Ντερούνεν. Ωστόσο, είναι δική μα αρμοδιότητα να συζητήσουμε αυτή την τεχνολογία ή μήπω πρέπει να το συζητήσει η αρμόδια επιτροπή. Ε, από εκεί και πέρα, για το πρώτο ερώτημα του κυρίου Άγγελ. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Θέλουμε πράγματι να φορολογήσουμε αυτές τις, να, μάλλον να απαγορεύσουμε αυτές τις ε, συναλλαγές τις χρηματιστηριακές που εκτιλήσονται μέσα σε νάνο δευτερόλεπτα και να τις απαγορεύσουμε στην Ευρώπη θα γίνονται παλού. Λοιπόν, εάν υπάρχει κάποια χώρα που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην Ευρώπη και έχει κάποιο σχέδιο διάσωσης, τότε ίσως υπάρξει κάποια διαδικασία προσωρινής ε, αναστολής αυτής της διαπραγμάτευσης, αυτού του είδους των ε, χρηματιστηριακών συναλλαγών, αυτού του είδους του trading δηλαδή. Τότε ε, θα μπορούσε κάποια συγκεκριμένη χώρα μόνο να το υιοθετήσει αυτό ως προσωρινό μέτρο. Και να δούμε και τα επιχειρήματα κατά αυτού του φόρου. Οι πράσινοι αναφέρθηκαν σε όλα αυτά άλλωστε. Το είπε και η κυρία Ντερούνεν. Πώς θα εμποδίσουμε να μετακυλιστεί ο φόρος αυτός στον καταναλωτή. Αλλά και τα ε, συνταξιδοτικά ταμεία ανησυχούν γιατί η θέσπιση αυτού του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών θα αυξήσει ε, το κόστος διαχείρισης των ε, χαρτοφυλακίων που διαθέτουν. Να εξετάσουμε και το θέμα από τη σκοπιά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ξέρετε, πολύ συχνά ε, λέγεται ότι οι μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις θα χάσουν. Δεν θα έχουν ε, οι τράπεζες χρήματα για να δανείσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εάν μειωθεί το περιθώριο ελιγμών που έχουν οι τράπεζες αυτή τη στιγμή. Αρχικά αυτός ο φόρος είχε παρουσιαστεί ως ο φόρος Τόμπιν, ο οποίος ε, είχε ως σκοπό να χρηματοδοτήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο παγκοσμίω. επομένως θα ήταν δύσκολο να πούμε ότι αυτή η ιδέα που έχουμε για το φόρο επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών θα εξυπηρετήσει το ίδιο, τον ίδιο σκοπό. Στην δική μου ομάδα οι απόψεις διήστανται, αλλά εγώ δεν θα ήμουν υπέρ της αυτόματης απόδοσης των εσόδων από αυτή τη φορολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον ευρωπαϊκό κορβανά. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να πάρουν τα χρήματα αυτά ε, τα κράτη-μέλη. Βέβαια, ε, αργότερα μπορούμε να δούμε αν τα χρήματα αυτά μπορούν να τύχουν κοινή χρήση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν θέλετε. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα το θεσπίσει αυτό το φόρο σε εθνικό επίπεδο στη Γαλλία. Τα ίδια παραδείγματα έχουμε και αλλού. Επομένως είναι αδύρυτη ανάγκη να προχωρήσουμε και από κάπου θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Ε, η χρηματοοικονομική κρίση προκλήθηκε εν από αυτές τις υπερταχείες συναλλαγές. Μπορούμε να περιμένουμε για μια πιο ευρεία συμφωνία βέβαια, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι θα επιτευχθεί ποτέ. Καλό θα ήταν κάποιος να ε, ξεκινήσει για να δώσει το καλό παράδειγμα. Ο Πρόεδρος, να πω και εγώ δύο λόγια από πλευράς της ομάδας μου γιατί ο σκιώδης εισηγητής δεν είναι εδώ και μάλλον τελικά μπορεί να καταλήξω εγώ να γίνω ο σκιώδης εισηγητής. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα εκπλαγείτε ακούγοντας ότι ε, ε, με πολύ σκεπτικισμό αντιμετωπίζω αυτό το ενδεχόμενο και χαίρομαι που ακούω ότι δεν είμαι μόνος. Να ξεκινήσω με μια γενική παρατήρηση. Έχω την αίσθηση ότι νομίζει ο κόσμος ότι είναι ένας εύκολος τρόπος ε, συγκέντρωσης κεφαλαίων ε, σε δυσμενείς συνθήκες για τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Μιλούμε για καινοτόμο χρηματοδοτικό μέσο, όσο αν μπορούσαμε να γεννήσουμε, αν θέλετε, έξτρα κονδύλια χωρίς να προκαλέσουμε ζημιά. Δεν εκπλήσωμαι καθόλου που ερμηνεύει την αξιολόγηση αντικτύπου διαφορετικά ο κύριος Σέμετα ε, με βάση, αν λάβουμε υπόψη μας, αυτά τα φρικτά οικονομικά στοιχεία που ε, ε, παρουσιάζονται εδώ και παραθέτω, λαμβάνοντας υπόψη το μετριαστικό αποτέλεσμα του σταθεροποιητικού μηχανισμού, το οποίο ήταν ε, απόν αν θέλετε, ο, ο αρνητικός αντίκτυπος εκτιμάται στο επίπεδο του μισού της εκατό. Τέλος της παράθεσης. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η αξιολόγηση αντικτύπου βρήθη επιφυλάξεων και νομίζω ότι ο αρνητικός αντικτύπος θα ξεπερνούσε κατά πολύ το μισό της εκατό. Λοιπόν, δεν θα πρέπει κατά την άποψή μου να υιοθετήσουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να μειώσει την ανάπτυξη του ΑΕΠ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να οδηγήσει σε ύφεση είτε μόνο κατά μισό της εκατό είτε και κατά πολύ περισσότερο. Ούτε έχουν αποδειχθεί τα, τόσο μεγάλα υποτίθεται ωφέλη του φόρου αυτού. Και υποτίθεται ότι θα έχει ε, αποτελέσματα προοδευτικά που θα διανέμονται προοδευτικά. Ε, είναι σαφές ότι πολλοί ε, που έχουν δουλέψει σε επιχειρήσεις για πάρα πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα βασίζονται στα συνταξιδοτικά προγράμματα των επιχειρήσεων αυτών. Και στη δική μου χώρα τα συνταξιδοτικά ταμεία επενδύουν σε μετοχές, σε ομόλογα, σε γραμμάτια ε, εθνικών κρατών, δημοσίου δηλαδή. Και περιμένουμε να υπάρχει σωστή διαχείριση χαρτοφυλακίου, πώληση, αγορά, μεταφορά των κεφαλαίων αυτών ε, σε μετοχές, σε ομόλογα, σε ομολογίες, ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη εγγύηση εξασφάλισης του κεφαλαίου. Και οι πολίτες βασίζονται σε αυτό. Πολλοί λοιπόν ε, πιστεύουν ότι θα περιοριστούν οι ικανότητες, όχι οι ικανότητες, οι δυνατότητες των διοικούντων τα, τα συνταξιωτικά ταμεία με τον φόρο αυτό. Δεν θα έχει ένα αποτέλεσμα με προοδευτική, αν θέλετε, κατανομή. Θα επηρεάσει όλους τους πολίτες, όλο το φάσμα της κοινωνίας και θα πρέπει η μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου να το λάβει υπόψη της αυτό. Τώρα, ως προς τον αντίκτυπο στον ε, χρηματιστηριακό ή χρηματοπιστωτικό κλάδο. Εν δυνάμει θα δημιουργηθούν προβλήματα στο, ε, στις αυτοματοποιημένες χρηματιστηριακές συναλλαγές. Έχω την αίσθηση ότι είναι μια πως στρεβλή πρακτική στις χρηματαγορές αυτή του αυτοματοποιημένου αν θέλετε trading αλλά αν τελικά αποδειχθεί ότι όντω είναι στρεβλή έχουμε και άλλους τρόπους να την αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε να ορίσουμε ποιες είναι οι αυτοματοποιημένες χρηματοστηριακές ε, συναλλαγές και να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό σε συνεργασία με τις αρμόδιες ε, ρυθμιστικές αρχές, επιτροπές κεφαλαγορών και το καθεξής ήδη σε αρκετές χώρες θα έχουμε επιπρόσθετη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, του χρηματοπιστωτικού κλάδου γενικότερα και αυτό δεν θα ευεργετήσει, δεν θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη. Οι τράπεζες νίζουν χρήματα στις επιχειρήσεις και μάλιστα σε επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Και το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν είναι σε θέση να το πράξουν αυτό, δεν το κάνουν αυτό, διότι έχουμε ε, βραδία ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να μην πω ύφεση. Και συμφωνώ βεβαίως με την κυρία Ρούνεν, περί τίνος πρόκειται άλλωστε. Η πρόταση αυτή θα δημιουργήσει ένα νέο διάβλο παραγωγής εσόδων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Κάτι το οποίο βεβαίως επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει κάτι στο οποίο ίδια θα έχει το first call αν θέλετε, στην οποία ίδια θα έχει τον πρώτο λόγο έσοδα που προκύπτουν από τον φόρο επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών μπορούν εν μέρη ή εις το όλο να αξιοποιηθούν για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Έτσι λέει το κείμενο, μόλις το παρέθεσα. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν η πρόταση αυτή δεν πείθη καθόλου και έχω την εντύπωση ότι δεν είναι καθόλου ρεαλιστική και δεν θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία εξουσία για να τα εξαναγκάσει να το κάνουν. Δεν πρόκειται να αποφασιστεί αυτό με τη διαδικασία της συναπόφασης. Δεν θα το δεχθεί η δική μου κυβέρνηση, αυτό είναι βέβαιο και πιστεύω και πολλές άλλες. Επομένως, θα προκληθεί μια στρέβλωση της εσωτερικής ενίας αγοράς. Και ο κύριος Άγγλ πρέπει να το πει αυτό στην έκθεση παραμένει αυτό το γεγονός ότι θα σημειωθεί μια κάποια στρέβλωση της αγοράς. Δηλαδή, οι χώρες που θα το θεσμίσουν θεσπίσουν αυτό το φόρο επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών θα χάσουν από πλευράς οικονομικής δραστηριότητας. Τώρα, αν ήταν αυτή η πρόταση μια συνολική, τότε θα είχε αξία να εφαρμοστεί ενδεχομένως αλλά από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί εν μέρη δεν θα λειτουργήσει και θα πλήξει τελικά τον Ευρωπαίο πολίτη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Αυτή λοιπόν ήταν η ε, συνεισφορά μου. Τώρα θα μιλήσω με την ιδιότητα του Πρόεδρου και θα πω ότι η κυρία Βανρόιτε και Γκέπχαρτ. Η κυρία Ρόιτόβα και μετά η εκπρόσωπος των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα δεν θέλω να επαναλάβω ότι έχει ήδη υποθεί στη συζήτηση αυτή. Ωστόσο, είναι μια συζήτηση που γίνεται στις χώρες μέλη και ειδικότερα στη δική μου χώρα, στην Τσεχία. Ε, τίθενται ξανά και ξανά τα ίδια ερωτήματα. Διότι δεν έχει σαφή στόχο η πρόταση αυτή τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να ρυθμίσουμε τον τομέα, θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό των κερδοσκοπικών ε, συναλλαγών ή μήπως θέλουμε απλά να ε, αποκτήσουμε περισσότερα εισοδήματα, έσοδα μάλλον φορολογικά, για να καλύψουμε συγκεκριμένες ανάγκες κοινωνικές. Αυτό είναι το ερώτημα. Τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Και δεν έχει καθόλου απαντηθεί. Από εκεί και πέρα, πού θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, πού θα αξιοποιηθούν ε, τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τη φορολόγηση αυτή. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευελπιστεί να ε, τύχει θετική αντίδραση η πρόταση αυτή από τα κράτη-μέλη, τότε θα πρέπει να τους πει ότι συμφωνεί ε, τα χρήματα αυτά να επιστρέψουν στον εθνικό κόρβανα, διότι αυτή τη στιγμή όλα τα κράτη προσπαθούν να βρουν τρόπους αύξησης των ε, εσόδων τους. Βεβαίως όλοι αντιλαμβανόμαστε τι προσπαθεί να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόταση αυτή. Ωστόσο δεν μπορούμε να είμαστε καθόλου βέβαιοι για το ποιο αντίκτυπο τελικά, ποιον αντίκτυπο θα έχει η πρόταση αυτή. Ε, ένα σωρό ερωτήματα ε, γύρονται για το τι θα γίνει εάν, εάν, εάν. Λοιπόν, είναι, χρειάζεται μάλλον μια πιο λεπτομερής ανάλυση και θα έλεγα επίσης ότι αφού είναι τόσο περίπλοκο το ζήτημα αυτό, θα ήταν καλό να οργανωθεί μια δημόσια ακρόαση ε, για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει τις διάφορες εναλλακτικέ οδούς με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μίας. Να παρουσιάσει δημοσίως τι μπορεί να επιτύχει ε, κάθε μία από τις διαθέσιμες επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Μιλώντα τώρα για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και ε, ο οποίος πολύ συχνά κατηγορείται ότι φέρει μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση, οφείλουμε να πούμε ότι ε, έχει μειωθεί η πιστοληπτική ικανότητα σε ορισμένες χώρες. Έχουν λάβει κάποιες χώρες μικρότερη βαθμολογία. Να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να φορολογήσει περισσότερο τα μερίσματα. θα πρέπει ενδεχομένω να εξεταστούν αυτά τα δύο θέματα, φορολόγηση μερισμάτων ή φορολόγηση χρηματιστηριακών συναλλαγών. Και τα δύο θα πρέπει να εξεταστούν. Ενδεχομένω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, θα έπρεπε να διερευνήσει περισσότερο ε, αυτές τις δύο επιλογές, αυτά τα δύο ενδεχόμενα. Και να ρωτήσω και τους συναδέλφους ποια είναι η γνώμη τους για τη δημόσια ακρόαση, για το ενδεχόμενο διοργάνωση δημόσιας ακρόασης για το θέμα αυτό. Επιτροπή σίγουρα ε, μπορεί να το κάνει, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο σε ό,τι αφορά τα θέματα ενιαία αγορά. Εάν δεν υπάρχει και χρόνο, θα δώσω τον το λόγο και δευτερολόγο. Θα δώσω λόγο στην συγκεκριμένη αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι πολύ περισσότερο χρόνο. Κύριε Καφαράτε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μου ξεφεύγουν ούτε και ξεχνάω τις τεχνικές δυσκολίες που υπάρχουν για τη δημιουργία ενός νέου εργαλείου, όπως ενός νέου, την εισαγωγή ενός νέου φορού για τις χρηματοπιστωτικές χρηματιστηριακές συναλλαγές. Κατ' εμέ όμως για να είναι, θα είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό όργανο για δύο λόγους. Το πρώτο αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το δεύτερο αφορά πιο συγκεκριμένα αυτό των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Είδαμε κάτι διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων ένα μέρος των δυσκολιών οι οποίες ε, έπληξαν τις χώρες μας. Και ένα μέρος επίσης των, των δυσκολιών που πλήττουν το ευρώ, που συνοδεύονται από μια χρηματιστηριακή ε, δραστηριότητα καθαρά κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ας μην μιλήσουμε για τις ε, εικονικές ε, μετοχές, ας μιλήσουμε για δράσεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένα στόχο να κερδοσκοπήσουν πάνω στην παρούσα χρηματοοικονομική κατάσταση μέσω ταχύτατων ανταλλαγών που δεν έχουν καμία άλλη αιτιολογία παρά μόνο να δώσουν πολύ μεγάλα κέρδη σε αυτός που τις πραγματοποιεί. Η πρακτική αυτή της ε, φύσης που είναι απόλυτα αρνητική απαιτεί να τύχει κάποιας, ε, κάποιες αντίδρασεις. Θα ήταν πραγματικά παράλογο να μείνουμε άπραγοι στην υφισάμενη κατάσταση θα ήταν πραγματικά παράλογο να απαντήσουμε ανταποκρινόμενοι και επανερχόμενοι δίνοντας συνθήκες οι οποίες προκάλεσαν αυτή την κρίση. Πρέπει πραγματικά να αποδυσαυρίσουμε την παρελθούσα εμπειρία και να προσπαθήσουμε να εισάγουμε νέα εργαλεία που θα διορθώνουν όλες αυτές τις αρνητικές συμπεριφορές, ξεκινώντας από αυτές των τραπεζών. Ένας φόρος λοιπόν που θα έχει σαν στόχο συγκεκριμένο την αποθάρρυνση των διαρθρωτικών δράσεων ουσιαστικά εξαιρετικά σημαίνει καθαρά συγκεκριμένου πολύ μικρού χρηματο, χρόνου επίδρασης θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη χρολόγηση ε, των δράσεων αυτών, αλλά και για το μήνυμα το οποίο θα στείλει ότι τέτοια είδου ε, κατάσταση, τέτοια είδου δράση δεν γίνεται πλέον ανοιχτή. Δεύτερο εξαιρετικά σημαντικό σημείο είναι αφορά την ε, προτινόμενη σχετική δράση του νομίσματος. Μιλάμε κατά κόρον για το τη σύμφωνα σταθερότητα και ανάπτυξη για να καταλήξουμε ότι κοιτάμε μόνο για σταθερότητα αλλά σχεδόν καμία ανάπτυξη. Πώ επιτυχάνεται η ανάπτυξη, απλά διευθετώντα του κανόνε τη αγορά, εγώ δεν το νομίζω. Η ανάπτυξη στην Ευρώπη έχει, είναι μονόδρομος με την κοινοτική δράση που θα πρέπει να αναλυφθεί. Γιατί καμία χώρα μόνη της δεν μπορεί να τα καταφέρει. Και με πολύ σημαντικές και γενναίες επενδύσεις στην κεντσιανή πολιτική η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή την ιστορική στιγμή στο σύνολο των κοινοτικών χωρών. Απαιτούνται λοιπόν πόροι. Μεμονωμένες οι χώρες δεν τις έχουν στη διάθεσή τους πόρους αυτούς. Αυτοί οι πόροι μπορούν να προκύψουν εν μέρη από το ευρωμόλογο εάν και όταν υλοποιηθεί, γιατί ενδεχομένως ένα μεγάλο ποσοστό μπορεί να χρησιμοποιηθεί των κονδυλίων αυτών για το ενιαίο ε, σύστημα ταμείο ε, αρρωγής και ένα άλλο κομμάτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επανακινήσει η οικονομία δεν θα έχει σχόλιο, θα λέτε και νόημα αυτό το δίλημα. Αυτή οι πόροι και αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να επαφηθούν στα, ε, στα κράτη-μέλη ή θα πρέπει να αποτελέσουν κομμάτι του προκοινωτικού προπολογισμού. Προφανώς το δεύτερο, σαν ένδειξη αλληλεγγύης. Νομίζω ότι σε συμπλήρωση όλου του διαρθρωτικού δίκτυου, του δίκτυου υποδομών που γίνονται στην κοινή αγορά, θα πρέπει να υπάρξει και σε αυτό το ιονί το εικονικό δίκτυο, για τα άειλα αγαθά. Ε, ζητώ συγγνώμη για την ειλικρίνη αυτή και την ομότητα, αλλά άκουσα να λέω ότι τα διάφορα τα, τα ταμεία ε, προνοίας μπορούν να, διαφυσβη, μπορούν να αμφισβητηθούν ή να διακινδυνεύσουν αν αναλάβουμε κάποια τέτοια δράση το αντίθετο. Εγώ θα έλεγα σε κανέναν να μην βάλει ευρώ, κανένα ευρώ σε αποταμίευση σε, μια, σε ένα ταμείο αλληλεγγύης, πρόνοιας, το οποίο πραγματικά δεν θα εγγυά τις συγκεκριμένε αποδόσεις και που δεν θα επιτηρείται σε κερδοσκοπικές πράξεις. Χρειαζόμαστε ακριβώς ταμεία τα οποία θα έχουν απόλυτη ασφάλεια, απόλυτη, ασφάλεια, απόλυτη σταθερότητα και θα εξασφαλίσουν με διαφάνεια τις αποταμιεύσεις μας. Τώρα, ε, είναι ή όλοι ή κανείς. Κοιτάξτε, το να υπάρξει μια συλλογική απαγόρευση σε οποιονδήποτε που για λόγους ακόμα και κατανοητούς, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, καθαρά εντός των εθνικών ορίων δεν θα πρέπει να λαμβάνεται κάποια δράση. Δεν, όταν λέμε ότι ό,τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος κάνει και η Ευρώπη, νομίζω ότι ουσιαστικά ψάχνουμε για δικαιολογίε και ε, δικαιολογίες. Εάν ξεκινήσουμε και δούμε ότι ο μηχανισμός λειτουργεί, θα είναι αρκετά εύκολο στη συνέχεια και άλλοι εκτός Ευρώπης που δεν είχαν πιστεί να μπορούσαν να ακολουθήσουν αυτή τη διαπρακτική. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό μπορεί να αντιπροσωπεύει πραγματικά ένα από τους πλέον καινοτόμους και ισχυρούς μηχανισμούς και ότι θα είναι θεμητό να χρησιμοποιηθεί προστασία σε ό,τι αφορά τον ορισμό του μηχανισμού και του ελέγχου. Και μπορεί να, δίνει, να κάνει και μια οριοθέτηση μεταξύ του πριν και του μετά. Επ' αυτού είμαι απόλυτα πεπισμένος για τη χρήση του νέου αυτού εργαλείου. Θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι έχουμε άλλο ένα σημείο στη μέση διάταξη να εξετάσουμε που είναι εξίσου σημαντικό. Και αυτό, κυρία Κέβερ, και νομίζω ότι και ο κύριος Βάρμπ ήθελε να λάβει το λόγο. Κύριος Βάρμπ. Η κυρία Σκάπα πρώτη. Δεν, δεν είμαι σίγουρος ότι έχω χρόνο για άλλον αγορητή. Κύριε Σκάπα. Η κυρία ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Άγγελ για την παρουσίαση. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια συζήτηση, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια πριν από λίγες καιρό ε, ζήτησε να εφαρμοστεί ο φόρος αυτός. Οπότε είναι λίγο παράξενο να ζητάμε το φόρο και μετά να ξαναρχόμαστε εδώ και να λέμε αν δεν ξέρουμε, δεν τον θέλουμε τώρα». Αυτό δεν είναι σωστό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ανταποκρίνεται θετικά σε ένα αίτημα του Κοινοβουλίου και κάνει αυτό που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επενείται. Δεν θα πρέπει να ε, φοβάται ότι θα αλλάξει γνώμη πάλι το Κοινοβούλιο. Και επίσης, εγώ βεβαίως έχω μία εντύπωση από την πρόταση αυτή, ότι είναι ένα είδος πλασίμπο η έκθεση, διότι δεν... Ε, ότι είναι απλώς ένα σκελετός χωρίς σάρκα και νομίζω ότι όπως είπε και ο κύριος Κορέα θα πρέπει να ε, δούμε στην πραγματικότητα τι πρέπει να κάνουμε και πώς μπορούμε να δώσουμε σάρκα και στην ε, πρόταση αυτή. Έχουμε πολλά να κερδίσουμε αν εφαρμόσουμε ορισμένα βασικά πράγματα. Δεν θα τα αναφέρω όλα αυτά, θα τονίσω ένα μόνο από αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Είμαστε πρώτα-πρώτα η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Και σε απάντηση σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Χάρμπορ εκ μέρους της πολιτικής του ομάδας. Πιστεύω ότι ή, ο φόρος αυτός μπορεί να είναι θετικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θα μας δώσει κάποια έσοδα με τα οποία μπορούμε να αναδιαρθρώσουμε και να μεταρρυθμίσουμε τη χρηματοπιστωτική αγορά Μπορούμε να φροντίσουμε να, ε, με αυτόν τον τρόπο να ωφεληθεί η πραγματική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να, για να οδηγηθούμε και σε ένα δίκαιο ανταγωνισμό Ο, γιατί όλα αυτά χρειάζονται χρήματα και αναχρηματοδότηση και όπως είπε και ο συνάδελφος Κομφεράτη για τα ταμεία συνταξιοδότησης. Υπάρχουν καλά ταμεία τα οποία δουλεύουν πολύ καλά και όπου οι πολίτες δεν χρειάζεται να φοβούνται ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα αλλά υπάρχουν και άλλα ταμεία τα οποία είναι ιδιαίτερα προβληματικά. Ακριβώς λοιπόν ε, να το να νοικοκυρέψουμε αυτόν τον τομέα, ακριβώ αυτόν τον τομέα, γιατί τι συντάξει παραδείγματο χάρη για τα συνταξιδοτικά ταμεία, είναι πολύ καλό για τον Ευρωπαίο πολίτη. Χρειαζόμαστε κάνουμε το νοικοκύρεμα αυτό. Αλλά ε, ε, μπορούμε μέσω αυτού του φόρου να βρούμε τα κονδύλια για να κάνουμε αυτό το νοικοκύραμα. Δεν πρέπει να βλέπουμε μοναχά τις αρνητικές πτυχές, πρέπει να βλέπουμε τις θετικές πτυχές της υπόθεση και να προσπαθήσουμε να τις αξιολογήσουμε και να τις χρηματο... και να τις ε, εκμεταλλευτούμε για ούτως ώστε να ε, επιδιώξουμε στόχους σε σχέση με την χρηματοπιστωτική αγορά που θέλουμε να ρυθμίσουμε καλύτερα. Σβάμπ. Αναρωτιέμαι, οφείλω να πω, κύριε Πρόεδρε, τι, κατά πόσο κατάλαβα καλά την επιχειρηματολογία α, ε, που ακούστηκε. Δεν πρόκειται για καινούριο φόρο εδώ δεν πρόκειται για έναν επιπλέον φόρο που δημιουργούμε ή που εμπνευστήκαμε για να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με πλέον έσοδα. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, τα συνταξιοδοτικά ταμεία δεν επηρεάζονται από το φόρο αυτό από το 0,01% που προβλέπεται για τις χρηματιστηριακές ε, συναλλαγές δεν κάνουν και τόσες πολλές. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο φόρος αυτός συζητιέται αυτή τη στιγμή γιατί θέλουμε κάποιους να τιμωρήσουμε. Ο Πρωθυπουργό του Ηνωμένου ε, Βασιλείου είπε ότι δεν μπορώ, θέλω να προστατεύσω το σύντη του Λονδίνου και δεν μπορώ να δοχθώ ορισμένα πράγματα. Και κάποιοι από τη Φραγκφούρτη λένε αντίστοιχα πράγματα. Σήμερα το πρωί μιλούσαμε για την Καλιφόρνια και λέγαμε ότι με τη ρύθμιση των σκαφών αναψυχής προχώρησε γρήγορα η Καλιφόρνια και έκανε ορισμένα πράγματα αρκετά νωρίς ε, και λέμε τώρα ξαφνικά ότι επειδή δεν θέλουμε στρέβλωση του ανταγωνισμού θέλουμε κι εμείς να κάνουμε ορισμένα πράγματα για τα σκάφια αναψυχής δηλαδή κάποιος άλλο το έκανε πρώτος και ακολουθούμε κι εμείς ε, Νομίζω λοιπόν ότι το πρώτο βασικό ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντήσουμε ως επιστροφή ε, ε, εσωτερικής αγοράς είναι το εξής. Γιατί μια εταιρεία όταν ε, κάνει κάποιες ε, ε επενδύσεις ε, ή επενδύει τέλος πάντων για κα, κάνει οποιασδήποτε επενδύσεις φορολογείται και γιατί δεν φορολογείται όταν αγοράζει μετοχές. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα δεν έχουμε πραγματικά χρόνο για, να, για δευτερολογία της Επιτροπής, αλλά αν θέλετε λίγο αργότερα, γιατί προφανώς ε, θα πρέπει να συνταχθεί και η γνωμοδότηση. Θα σας προσκαλήσω λοιπόν να ξανάρθετε όταν ο κ. Έντουιν καταλήξει. Ελπίζω να μπορέσει να κάνει, να κάνει κάποια λογική πρόταση, να αποσαφινιστούν τα πράγματα. Θέλετε να ακούσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ναι, ξέρετε ότι έχουμε μόνο μία ώρα για την παρουσίαση. Και υπάρχει και ένα ακόμα θέμα πρωτού ξεκινήσουν οι συντονιστέ. Λοιπόν, θα έχει την ευκαιρία να ακούσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνέχεια τον κύριο Άγγελ θα έχει ετοιμάσει τι ιδέε του. Ναι, πάρτε το λόγο, ναι. Κατανοώ του ε, χρονικού περιορισμού, αλλά θα ήταν ίσω ενδιαφέρον και σε σχέση με αυτά που ελέγχθησαν από ήδη προηγουμένω, τι έχει να μα πει η Επιτροπή σε σχέση με μια δεύτερη ή αναθεωρημένη ή μια τελείως καινούρια ε, μελέτη επιπτώσεων. Ευχαριστούμε πολύ. Η αναθεωρημενη η μια τελειως καινουρια μελετη μπορεί να μας μιλήσει περί αυτού. Κύριε Ντιμά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα να παρέμβω σε πάρα πολλά θέματα, αλλά θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Λίγα σημεία. Δεν θα υπάρξει αναθεωρημένη ε, μελέτη αντικτύπου. Αυτό το οποίο έκανε η Επιτροπή και τώρα είναι στην τελική της ε, τελειοποίηση είναι σχετικές ασκήσεις προσωμείωσης του χρηματοοικονομικού αντίκτυπου που θα μπορούσε να προκύψει από την εφαρμογή της πρότασης αυτής. Και αυτό δεν είναι προκειμένου να παίξουμε και να αποφύγουμε διάφορα παίζοντα με τα νούμερα όπω υπονοείται, υπονοείτε, αλλά γιατί η μελέτη αντίκτυπου έγινε το πρώτο εξάμεινο πέρσι ήταν γενική υφή. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να στοχεύουμε πιο συγκεκριμένα στι ασκήσει προσωμείωση που έχουν γίνει πάνω στι ε, συγκεκριμένε λεπτομέρειε της πρότασης που σας έχει υποβληθεί προς εξέταση. Και πλέον τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία τα οποία ε, μελετώνται τώρα είναι πολύ πιο καλά αν θέλετε. Φαίνεται ότι η απώλεια του ΑΕΠ, ε, επενδύσεις, απασχόληση, κεφαλογικό κόστος επενδύσεων κλπ είναι ουσιαστικά σχεδόν αγνοούμενες οι επιπτώσεις μακροπρόθεσμα από την επιβολή ενός τέτοιου φόρου. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα. Σε κάθε περίπτωση, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαμε να διτάξουμε ότι μια οποιαδήποτε μελέτη αντίκτυπου θα έδειχνε κάποια αρνητικά χρηματοοικονομικά συμπεράσματα, δεν θα κατέληγε, αν θέλετε, συμπερασματικά ε, στο εναντίον της πρότασή μας. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η έκθεση αντίκτυπου. Είναι δηλαδή μια εκ των προτέρων μοντελοποίηση του αντίκτυπου. Δεν, δεν γίνεται τίποτα, καμία χρήση ό,τι αφορά τον ορισμό και τη χρήση του εισοδήματος. Υπάρχουν κάποιοι ορισμοί του χρηματοοικονομικών συναλλαγών που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε οικονομικό μοντέλο κλπ. κλπ. Αν μου επιτρέπετε εντάχει, ένα σημείο το οποίο ε, επανήλθε στις ε, παρεμβάσεις πολλών από τους βουλευτές και που είναι σημασία στην Επιτροπή αυτή είναι ο αντίκτυπος στην εσωτερική αγορά. Στη θεωρητική περίπτωση που κάποια υποομάδα κρατών μελών εφάρμοζε τον τάξη και όχι, τον, το φόρο αυτό και όχι το σύνολο των 27 χωρών. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει μια πρόταση για το σύνολο των κρατών της Ευρωπαϊκής Εάν υπήρχε μια τέτοια εξέλιξη πρωτοβουλία με κρατών μελών και όχι από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσουν σε εφαρμογή σε ένα υποσύνολο κρατών, θα υπέθετε ότι αυτό θα γινόταν μέσω του, ε, ε, μέσω του μηχανισμού ενισχυμένης συνεργασίας που προβλέπεται από τι ευρωπαϊκέ συνθήκε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ελέγξει κατά πόσον υπάρχει αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά που ενδεχομένως θα έκανε αδύνατη την εισαγωγή ενός τέτοιου ε, φόρου σε κάποιες λίγες χώρες μονοκράτες μέλη. Δεν μπορώ να προδικάσω το αποτέλεσμα, αλλά σκεφτείτε όπως στο ΦΠΑ, όπου έχουμε υφιστάμενο πλαίσιο κοινοτικών νόμων σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ, με διαφορετικούς ΦΠΑ σε διάφορες χώρες, αλλά θα ήταν δύσκολο να δούμε. Για παράδειγμα, τη φορολόγηση αυτοκινήτων. Εάν δεν υπήρχε αυτή η ενιαία προσέγγιση, δεν θα οδηγούσε τι απαραίτητε αλλαγέ σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεν μπορώ λοιπόν να προδικάσω τι αξιολογήσει αυτέ, αλλά πάντως θα γίνει και ίσω εξίσου σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι υπάρχουν και υποχρεώσει μη επιβολή αρνητικών διακρίσεων ε, και του κοινοτικού νόμου έναντι των τρίτων χωρών που την άποψή μα δεν παραβιάζεται από την τρέχουσα πρόταση και θα μπορούσε να μα δώσει μια περαιτέρω ένδειξη του τι θα μπορούσε να συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν μόνο μια υπομάδα κρατών προχωρούσε. Αλλά βέβαια είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναλυθεί λεπτομερώς και εν ευθέτω χρόνο εάν και όποτε ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία. Έχοντας επίγνωση της ε, στενότητας χρόνου, σταματώ εδώ, αλλά βέβαια είμαι στη διάθεσή για οποιαδήποτε τεχνική συμφίση ερωτήματα θέλετε να υποβάλλετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ανταποκρινόμουν στο τελευταίο ερώτημα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το πότε, όχι το εάν. Προτείνω λοιπόν αρχίστε να δουλεύετε άμεσα για την εφαρμογή του φόρου αυτού νωρίτερα. Γιατί πιθανότατα η δική μου χώρα μάλλον δεν πρόκειται να αλλάξει άποψη. Αν στοιχημάζα λοιπόν θα έλεγα ότι εκεί ακριβώς πρέπει να επικεντρώσετε τις προσπάθειές σας. Κύριε Άγγελτ, έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα εδώ. Θέλετε να τίποτα περισσότερο? Θα μας στείλετε το προσχέδιο της έκθεσης τέλη Φεβρουαρίου ή κάνω λάθος. Είχα την πρόθεση να είμαι λίγο νωρίτερα. Εν πάση σίγουρα μέχρι τις τέλος Φεβρουαρίου θα το έχετε την έκθεση. Δεν ξέρω ποια θα είναι η αρχική γλώσσα σύνταξης της έκθεσης. Ενδεχομένως να είναι επίσης αγγλικά δεδομένου ότι τα πράγματα έχουν, όπως έχουν κινηθεί τα πράγματα μέχρι στιγμή, και όπως πολύ σωστά είπατε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τα θέματα εσωτερική αγορά και τη εφαρμογή από χθε. Και αυτό σκοπεύω να κάνω στην πρόταση που σκοπεύω να υποβάλλω για επιζητώντα βέβαια την προσοχή σα και ζητώντα την υποστήριξή σα. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζουμε ότι ήταν πολύ σημαντική και επικοδομητική συζήτηση και προσβλέπουμε στη τελική σα έκθεση για να συνεχίσει η συζήτηση. Προχωράμε λοιπόν σε αυτό που πιστεύω ότι θα είναι μάλλον σύντομο, αλλά αρκετά σημαντικό, γιατί πρέπει να παρακολουθήσουμε και κάποιες αλλαγές. Διότι, όπως ξέρετε, στην, ως τμήμα της προκαταρκτικής εργασίας μας στην, έκθεση εφαρμογής στην ε, οδηγία καταναλωτικής πίστης ε, ε, παραγγείλαμε κάποια μελέτη η οποία έγινε από το Ινστιτούτο Νομικών ε, υποθέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνδεση με κάποιο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Έχετε ένα αντίγραφο λοιπόν στο πακέτο σας. Και νομίζω ότι και ευχαριστώ και το τμήμα εκπόνησης πολιτικής που μας είναι γνωστό και που έχει προετοιμάσει σχετική μελέτη για μας. Δυστυχώς ο κύριος Τσόλ από το Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας που ήταν επικεφαλής ε, έχει αποκλειστεί λόγω χιονιού στο Μόναχο. Όσοι σκοπεύουν να επιστρέψει την Παυαρία, πρέπει να το ξέρετε. Αλλά η κυρία Μαργαρίτα Λαβίνοβιτς από το Πανεπιστήμιο του Βόσεμπουργκ επίσης ε, έχει, είναι εκτός. Έχω την μελέτη σας και το ε, βιογραφικό σας εδώ στα γερμανικά, τα αγγλικά αλλά και την Πολωνία. Θα μας παρουσιάσει λοιπόν τη μελέτη, είναι εδώ ευτυχώς, και θα μας παρουσιάσει τη μελέτη εκ μέρους της. Εάν είναι δυνατόν να το κάνετε μέσα σε ένα δεκάλεπτο, ώστε να έχουμε και λίγο χρόνο για συζήτηση. Και φοβάμαι ότι και ο κύριος Λέχνα έχει καθυστερήσει λόγω τρομερούς διαλόγου και ελπίζουμε αν καταφέρει να ολοκληρώσει συζητήσει εγκαίρως να έρθει. Ε, Ταξί προτείνω σε οποιοδήποτε συνέχεια να παρουσιάσει τις προτάσεις. Θα ακούσουμε πρώτα τη μελέτη από την κυρία Λαβίνοβιτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Μας ανησυχεί η εφαρμογή της οδηγίας περί καταναλωτικής πίστης σε μας το Ινστιτούτο θα σας παρουσιάσω μερικές, θα σας δώσω μερικές γενικές ε, πληροφορίες για τη μελέτη, κάποιες γενικές παρατηρήσεις σχετικά με την τυπική εφαρμογή της οδηγίας και προσπαθήσω να, κάνω, να αναλύσω ορισμένες τυχές της οδηγίας και τελικά θα μιλήσω και για την ε, διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Κοιτάξτε, το Προσπαθήσαμε να μελετήσουμε τις κύριες δυσκολίες στην εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Πρόκειται για μια οδηγία πλήρους εναρμόνισης. Αυτό δημιουργεί δυσκολίες. Βεβαίως για ορισμένα σημεία υπάρχει περιθώριο ελιγμών, θα τα δούμε και αυτά. Και μετά θα μιλήσουμε και για τις τις εναλλακτικέ λύσεις που αναφέρονται, που μπορεί κανείς να επιλέξει, τις επιλογές που έχει κανείς και που αναφέρονται στην οδηγία. Και για κάποια σημεία της οδηγίας που απαιτούν περαιτέρω εξηγήσει. Η μεθοδολογία μας ποια ήταν. 14 κρατη μέρια μελετήσαμε Έχουμε στοιχεία από 14 κράτη-μέλη δηλαδή. Τα επιλέξαμε πώς. Προσπαθήσαμε να έχουμε κράτη-μέλη και εθνικού δικαίου και ε, ρωμαϊκού δικαίου και καινούριε χώρες και παλιές χώρες και βεβαίως όλα τα κράτη-μέλη με τα οποία ασχοληθήκαμε ε, έχουν εφαρμόσει την οδηγία έξι εξ αυτών καθυστερημένα. Είπαν Ε, έδωσαν αυτά τα έξι κράτη-μέλη δικαιολογίες για το γιατί καθυστέρησαν στην εφαρμογή ε, ποια ήταν τα εμπόδια που αντιμετώπισαν. Σε αντίθεση με την πρώτη οδηγία του 1987, η οδηγία αυτή προβλέπει πλήρη εναρμόνιση. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη διατηρούν, εισάγουν νέες νομοθετικές διατάξεις, αλλά δεν επιτρέπεται να ξεπεράσουν καθόλου το επίπεδο προστασίας που προβλέπεται. Αυτά είναι τα ε, σημεία για, τις, ε, στα οποία, ε, για τα οποία υπάρχουν διατάξεις πλήρους εναρμόνισης Έχουμε το ΣΕΚΙ, έχουμε το περιεχόμενο της σύμβασης, έχουμε το δικαίωμα ε, επαναχώρησης, ε, δυνατότητες ε, πρώιμης, ε, ε, αποπληρωμής κτλ. Λοιπόν, για το ΣΕΚΙ, έξι από τα 14 κράτη-μέλη εφάρμοζαν ακριβώς την οδηγία τέσσερις, τέσσερα κράτη-μέλη άλλαξαν ε, λιγάκι τη διατύπωση αλλά ελάχιστα το περιεχόμενο ήταν το ίδιο αλλά τε, τέσσερις χώρες εφάρμοσαν με κάποιες αλλαγές ακόμη και στο περιεχόμενο και επί της ουσίας της οδηγίας δηλαδή παράδειγμα ε, η Γαλλία δεν εφάρμοσε τα του δικαιώματος ενημέρωσης. Η Πορτογαλία για την δεν εφάρμοσε το κομμάτι για την προειδοποίηση σε περίπτωση ε, ε, πρόορης αποπληρωμής. Τώρα, Thank you. Um, we Τώρα το δεύτερο σημείο που ανέφερα είναι το περιεχόμενο της σύμβασης. Αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα, μόνο η Ρουμανία και η Λετωνία. Ε, δεν εφάρμοσαν ένα κομμάτι τε, του το σημείο 15 στη Γερμανία η μεταφορά ήταν σωστή αλλά συμπεριέλαβε και επιπλέον κυρώσεις για το 14.1β. Τώρα για το δικαίωμα υπαναχώρησης που είναι το τρίτο θέμα που, για το οποίο θα ήθελα να σας μιλήσω. Όλα τα κράτη-μέλη το εφάρμοσαν αυτό, αλλά φαίνεται ότι το δικαίωμα αυτό δημιουργήσε τα μεγαλύτερα προβλήματα στα κράτη-μέλη. Λόγω χάρη στη Γερμανία υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψει επιστροφής. Εκείνη είναι εναλλακτική λύση σε σχέση με την υπαναχώρηση αυτή. Ε, αυτό ίσως δεν είναι πλήρως μέσα στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία δεν είναι έννοια τη πλήρου Τελικά, με την, σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή, δεν υπήρχαν προβλήματα, αλλά υπήρχαν αρκετές επικρίσεις και όπως ήδη είπα η Πορτογαλία ε, εισήγαγε μια νέα διάταξη για την υποχρέωση προειδοποίησης σχετικά 30 μέρες πριν από την δυνατότητα του πελάτη να αποπληρώσει οποιοδήποτε δάνειο. Τώρα, μια και δεν έχουμε χρόνο να αναφερθώ στις διατάξεις που μπορούν να ερμηνευτούν με τις ευρείες διατάξεις μπορούν να ερμηνευτούν με διαφορετικούς τρόπους. Άρθρο 5 παράγραφος 6 αναφέρεται στο περιθώριο εκτίμησης. και το 15.2 για τις, ε, ε, τις αποζημιώσεις ας πούμε και ή αντιθέτω κυρώσει. Το άρθρο 6 εφαρμόστηκε από όλα τα κράτη-μέλη, 9 των κρατών μελών. Parameters which are not Ε, έκανε κάποιες, δεν έκανε ορισμένα, δεν εφάρμοσαν πλήρως Ε, οι Γερμανοί ήταν αυστηροί όσον αφορά τι εξηγήσει πρέπει να δίνονται για την κατανόηση του σύμβαση από τον καταναλωτή. Excuse me. Um, the second part is the margin of appreciation as regards the, ex, um, the extent to, the, to which το επόμενο θέμα είναι, σχετίζεται με το άρθρο 15 γιατί για τις αποζημιώσεις αν μπορούμε να το πούμε έτσι ή τις κυρώσεις κάποιες χώρες έκαναν μικρές αλλαγές εδώ η Γερμανία δεν διατήρησε τον δευτερεύοντα χαρακτήρα της διάταξης. Όσον αφορά τις κυρώσεις, περισσότερες χώρες εφάρμοσαν τα σχετικά σωστά. Είναι ε, κυρώσεις αστικού, αστικές, αστικού δικαίου οι περισσότερες από αυτές που τα πρόστιμα ας πούμε που επιβάλλονται εδώ. Θα μπορούσαμε... Τώρα έρχομαι στις επιλογές που, για τις οποίες δίνει δυνατότητα η οδηγία. Η Βουλγαρία δεν επέλεξε καμία επιλογή. Η Αυστρία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία μία επιλογή. Η Κύπρος, η Ρουμανία επέλεξαν τις περισσότερες επιλογές. Από τις επιλογές η, αυτή του άρθρου 2.6 επελέγει από τους περισσότερους γιατί και η επιλογή του άρθρου 16.4 ήταν επίσης αρκετά δημοφιλής. για την πρόορη αποπληρωμή και την αποζημίωση η οποία είναι περιορισμένη σε αυτή τη δυνατότητα. Οι επιλογές που δεν επελέγησαν ήταν αυτές που σχετίζονταν με την μείωση, αν θέλετε, από μείωση του δικαιώματος υπαναχώρησης ή ε, ε, αυτές που ε, προβλέπουν μεγαλύτερη αποζημίωση. Τα κράτη-μέλη λοιπόν σε γενικέ γραμμέ εμεί πιστεύουμε ότι επέλεξαν δυνατότητε που του δίνεται από τη οδηγία που είναι υπέρ του καταναλωτή. η επιλογές που έγιναν από τα κράτη-μέλη ε, δεν σχετίζονται με το χρόνο ε, μέσα στον οποίο εφάρμοσε το κράτος μέλος αν εφάρμοσε νωρίς ή αργά αν θέλετε τώρα για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής 9 από τα 14 κράτη-μέλη διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής και εφαρμόζεται η οδηγία και σε δεύτερες υποθήκες όπου δίνονται κάποια δάνεια ας πούμε για να... και σε γενικές γραμμές ε, αυτά εφαρμόζονται ιδιαίτερα ε, για τη χρηματοδότηση ακινήτων. Ναι, θα ήθελα να δείτε και το πίνακα που έχουμε στο τέλος του, της μελέτης να, θα έλεγα να τον δείτε για την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα αυτό. Είναι πολύ πιο εύκολο να το παρακολουθήσω διαβάζοντας την έκθεση παρά κοιτάζοντας τη διαφάνεια, οφείλω να πω. Ο κύριος ε, Λέντινορ είναι εδώ, κατάφερε να ξεγλιστρήσει από τον τριμερή ε, διάλογο στον οποίο ε, συμμετέχει. Θέλετε να πάρετε το λόγο, να σχολιάσετε τα λεχθέντα, τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί δεν μπορούμε φυσικά να προχωρήσουμε σήμερα το απόγευμα. Νομίζω ότι πρέπει να το διαβάσουμε, να διαβάσουμε την έκθεση προσεκτικά και να το συζητήσουμε σε επόμενη συνάντηση. Αλλά πείτε μας κι εσείς ε, την άποψή σας. Ευχαριστώ πολύ πρώτα πρώτα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί έλαβα μέρος σε δύο τριμερείς διαλόγους. Ο πρώτος ήταν ε, επιτυχής, ο δεύτερος δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ήταν πάρα πολύ δύσκολη η διάλογη αυτή ε, όσον αφορά το αντικείμενο ε, της, του, του διαλόγου. Το Ηνωμένο Βασίλειο, κύριε Πρόεδρε, έχει μεγάλη σημασία, αλλά είναι δύσκολος συνομιλητής. Τέλος πάντων το δεύτερο διάλογο τον διακόψαμε πιο νωρίς το πράγμα που με βόλευε εμένα γι' αυτό βρίσκομαι εδώ αλλά επιπλέον ήταν αναγκαστικό γιατί δεν προχωρούσαν τα πράγματα. Λοιπόν, για την οδηγία που συζητούμε εδώ περί καταναλωτικής πίστης. Προσπάθησα να, να δω πώς εφαρμόζονται ορισμένα πράγματα στη χώρα μου. Πριν από ένα-δυο χρόνια α, το, το μελέτησα για πρώτη φορά αυτό, να δω πώς εφαρμόζεται η οδηγία δηλαδή στη Γερμανία. Εν τω μεταξύ ξέχασα και τα συμπεράσματά μου, αλλά τώρα βεβαίως έχουμε μια επίσημη μελέτη η οποία αναφέρεται στο το ότι έκανα περισσότερα από ένα κράτος μέλος και από τη μελέτη αυτή φαίνεται ότι πολλά κράτη-μέλη εφαρμόζουν την οδηγία αυτή στα ενυπόθηκα δάνεια τα οποία δίνονται κτλ. Αυτό το περιμέναμε. Δεν θέλουμε Χαιρόμαστε που εφαρμόζονται, εφαρμόζονται οι οδηγία αυτοί Δεν χρειάζεται να κάνουμε καινούργια οδηγία βέβαια που να λέει το αντίθετο από αυτά που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή. Ε, πολλά πράγματα έχουν ρυθμιστεί, αλλά πρόκειται για περίπλοκα πράγματα. Παραδείγματο χάνει το δικαίωμα προώρη αποπληρωμή. Ε, είναι περίπλοκο. Συνήθως η καταναλωτική πίστη, τα δάνεια, τα καταναλωτικά που δίνονται είναι μικρή χρονική διάρκεια. Δεν είναι σαν τα ενυπόθηκα δάνεια. Οπότε ε, ε άλλα πράγματα ισχύουν για την πρόορια αποπληρωμή για ενυπόθηκα δάνεια πριν μεγάλες διάρκειες και άλλα εδώ για ε, βράχη πρόθεσμα αν θέλετε καταναλωτικά δάνεια. Ε, ε, εκείνο που θα ήταν ενδιαφέρον θα ήταν να δούμε βέβαια τα επιτόκια α, ε, που εφαρμόζονται, ποια είναι, αν είναι ομοιόμορφα ή αν τέλος πάντων αν μοιάζουν εκεί που στις διάφορες χώρες γιατί αυτή είναι η καθημερινότητα ε. Ε, θα πρέπει να τη δούμε λοιπόν τι είναι τα επιτόκια και να δούμε μετά και σε ε, τρία-τέσσερα χρόνια ε, τι γίνεται με τα δάνεια αυτά, τα διασυνοριακά ιδιαίτερα δάνεια που μπορεί να πάρει ένας καταναλωτής που ζει σε μια χώρα από μια άλλη χώρα. Ε, βεβαίως, ε, να σας πω τώρα κλείνοντας ότι φεύγω, ότι κλείνει, τελειώνει στα διοδρομία μου, θέλετε, εδώ στο, στο Κοινοβούλιο, στις 17 Μαρτίου ε, φεύγω ε, και η διάδοχος μου βεβαίω είναι μια κυρία η οποία, η οποία είναι νομικός ε, και η οποία εισάξια θα με εκπροσωπήσει, θα με διαδεχθεί βεβαίω. αλλά επειδή ακριβώς φεύγω στις 17 Μαρτίου θα πρέπει να δούμε ακριβώς το χρονοδιάγραμμα και η της, για την έκθεση αυτή τι θα είναι, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα πιο εκπληκτικά νέα που ακούμε σήμερα το απόγευμα, ότι θα αποσυρθείτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Ήσασταν, ε, είσαστε ένα από τα μέλη που έχουν υπηρετήσει περισσότερο ε, το θεσμικό αυτό όργανο και με τον καλύτερο τρόπο. Σας ευχόμαστε το καλύτερο. Είναι θέμα που θα πρέπει να εξετάσουν τους συντονιστές, οι συντονιστές. Και βεβαίως η, η χρονική συγκυρία πρέπει να εξεταστεί, το χρονοδιάγραμμα πρέπει να εξεταστεί. Να δούμε πώς θα ταιριάξει η δουλειά αυτή με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπω και την κυρία Ρούσο, η οποία ήρθε για να ακούσει για τα θέματα αυτά, γιατί θα, τα, θα δουλέψει πάνω σε αυτά τα θέματα ε, από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Να συζητήσουμε λοιπόν το χρονοδιάγραμμα με την Επιτροπή και ο κύριος ΦΑΜ να ε, δώσει μια αναφορά στους συντονιστές. Να ευθυγραμμίσουμε δηλαδή τη δουλειά μας μεταξύ μας. Να έχουμε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε πολιτικά ε, ως προς αυτή την πολύ σημαντική οδηγία για να μπορέσει να λάβει υπόψη της τις απο σύμβης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Αυτή είναι η πρότασή μου, εάν συμφωνούν και οι άλλοι συντονιστές. Επομένως, ο κύριος Πουσόλη είναι εδώ, είναι και εκείνος σκιώδης εισηγητής. Προτείνω λοιπόν να κλείσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό στο σημείο αυτό σήμερα το απόγευμα να ευχαριστήσουμε την κυρία Λαβίνοβιτς, ζητώ συγγνώμη αν δεν προφέρω σωστά το όνομά σας, να πάρουμε λίγο χρόνο να χωνέψουμε αυτή την έκθεση, να διαβάσουμε καλύτερα ε, τα στοιχεία και τα νούμερα και στη συνέχεια να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα συζητήσουμε για το χρονοδιάγραμμα κτλ. Συμφωνείτε όλοι? Καλώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Επομένως, ε, ολοκληρώνω τη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, σήμερα το απόγευμα εδώ. Αύριο το πρωί θα τα πούμε στις 9. Θα έχουμε παρουσίαση της Δανέζικης Προεδρίας. Θα ακούσουμε το Δανό Υπουργό για τις Επιχειρήσεις και την Απασχόληση, τον κύριο Όλι Ζών, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα τριών λεπτών μέχρι να αποχωρήσουν όλοι από την αίθουσα και στη συνέχεια θα λάβει χώρα η συνεδρία των συντονιστών. Ευχαριστώ.